That we have... Ε, γεια σας. Ε, λοιπόν, ας αρχίσουμε ε, να διεκπαιρώσουμε μερικά πράγματα πριν έρθει ο Επίτροπος. Διερμηνέα έχουμε σε όλες τις γλώσσες εκτός από μαλτεζικά, κροατικά, λετονικά και ρουμανικά. Δεύτερο σημείο, αναφορά από την ε, επίσκεψη αντιπροσωπεία ΕΜΠΕΛ στο κόμμα και το Ρήνο 29 με 31 Οκτωβρίου του 2018. Θα βρείτε την έκθεση στα ε, εγγραφά της συνεδρίασης. Σημείο 3 αναφορά από τις ε, τρέχουσες δια, οργανικές διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Κώσα θέλει να μας ενημερώσει πάρα πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια πολύ ιδιάζουσα κατάσταση και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους διότι Κανονικά θα έπρεπε να σας είχα ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα, αλλά είχε καθυστέρηση η πτήση μου, οπότε θα το κάνω τώρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα των συζητήσεων και την οδηγία ε, για την προσβασιμότητα. Όπως γνωρίζετε το 2015 κατέθεσε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάστηκε μια τριετία εργασιών για να ολοκληρωθούν και να κλείσουν οι διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω την άλλη εβδομάδα, στις 19 του μηνός θα αποφασίσει η Κορεπέρ για αυτά τα θέματα, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και μάλλον θα υποστηρίξει την πρόταση. Στο Κοινοβούλιο η Επιτροπή Οικοσυτερικής Αγοράς θα ψηφίσει στις 22 ε, Ιανουαρίου και το Μάρτιο θα πάει στην Ολομέλη. Τέσσερα είναι τα βασικά αποτελέσματα που θα πρέπει να σας ενημερώσουμε γι' αυτά. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχουμε το τελικό ε, κείμενο. Ε, τρέχουν ακόμα οι ε, διαπραγματεύσεις. Η οδηγία θα επιτρέπει και στους παρόχους υπηρεσιών αλλά και σε κατασκευαστές προϊόντων να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες και έτσι οι καταναλωτές με αναπηρία ε, θα έχουν μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων όσο και υπηρεσιών στη διάθεσή τους. Είναι πολύ καλό ε, υπάρχουν ε, τερματικοί στάθμοι για πληρωμές, για ε, self-service ε, με τα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, πρόνοια για τον τουρισμό, ακόμα και το 112, αυτό το τηλεφωνικό νούμερο είναι τώρα πλέον υποχρεωτικό να υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη και με πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία. Ε, σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις μέχρι και διαφωνίες. Τα κράτη-μέλη δέχτηκαν την εθελοντική προσέγγιση. Βλέπω έφτασε η Επίτροπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέλαβε να βολιδοσκοπήσει τα κράτη-μέλη και να μας ενημερώσει ε, σχετικά με αυτή την εθελοντική προσέγγιση που επελέγει τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, μετά από μία τριετία έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση, μεγάλη πρόοδος και οικονομική και κοινωνική. Θελήσαμε περισσότερα βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις να επιτύχουμε, αλλά θέλαμε και να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για να τελειώσουμε και να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Για να μην υπάρξουν λοιπόν και άλλες καθυστερήσεις, συμφωνήσαμε. Ευχαριστώ κύριε Κώσα. Όλοι γνωρίζουμε ότι συνεχίζονται ακόμα οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και σε πολλά θέματα, καθώς ε, τελειώνει η θητεία μας, θα επανέλθουμε σε αυτά, όχι σήμερα. έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και να κλείσουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα πριν ε, εκπνεύσει η θητή. Θέλει να πει τίποτα ο κύριος Κάσα, όχι. Προχωρούμε λοιπόν. Στην έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων. Καλώς ορίζουμε την Επίτροπο κυρία Τέσεν. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Έρχεστε στην Επιτροπή κάθε φορά που σας καλούμε και άλλες φορές μας τηλεφωνείτε εσείς και μας λέτε να έρθω να σας ενημερώσω στην Επιτροπή. Και τώρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, βρίσκεστε εδώ για να μας παρουσιάσετε την ετήσια ε, μελέτη για την ανάπτυξη για το 2019 και θα σας δώσω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα, από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ε, ε, παρουσιάσω αυτή τη δέσμη ε, του φθινοπορεινού εξαμήνου 2019, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το σχέδιο έκθεσης για την απασχόληση. Η Ευρώπη ε, βρίσκεται σε φάση οικονομικής ε, μεγέθησης, ανάπτυξης. Ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν και ε, γερή, στιβαρή, υγιή. Εν πάση περιπτώσει, μετά από έξι χρόνια διάλειπτης οικονομικής μεγέθυνσης έχουμε μείωση της ανεργίας και ανάπτυξη ακόμα και σε χώρες που έχουν χαμηλότερο κατακεφαλή ΑΕΠ. Πάνω από 239.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά. Ε, ο δείκτης απασχόλησης πλέον είναι στο 73% και μπορούμε να ε, πούμε ότι φτάνουμε κοντά στο στόχο της Ευρώπης 2020 ε, που είναι 75% μέχρι το 2020. Έχουμε θετικά και στην κοινωνική πολιτική είναι λιγότεροι φτωχοί και αποκλεισμένοι. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα πριν της κρίσης. Μόλις πέρσι 5 εκατομμύρια, ή μόνο πέρσι 5 εκατομμύρια ε, πολίτες βγήκαν από τη φτώχεια ή από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τελικά υπάρχει κάποια πρόοδος ε, συγκρατημένη, δεν υπερβάλλω, προς τους στόχους 2020 για την ε, αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού. Πραγματικά κάνουμε πρόοδος και είναι σημαντικό διότι ε, βλέπουμε και την τάση να συνεχίζεται και το 2019 και αυτό είναι πολύ ε, ενθαρρυντικό. Το κοινωνικό βαθμολόγιο, τι είναι αυτό, είναι κάτι που συνοδεύει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ήδη από πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχουμε εντάξει ε, αυτό το δίκτυο και για δεύτερη φορά στην κοινή έκθεση και μάλιστα με πλήρη τρόπο. Ε, ε, Πέρυσι είχαμε 12 από 14 δείκτες, τώρα έχουμε και τους 14. Και τι μάθαμε από τα αποτελέσματα αυτού του κοινωνικού βαθμολογίου. Έχουμε παντού βελτίωση σε 13 από 14 δείκτες τίτλους. Με εξαίρεση την επίπτωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων για τη μείωση της φτώχειας που έχει πέσει και έχουμε και τον αυτόματο σταθεροποιητή σε περίπτωση οικονομικής ε, ανάπτυξης και επέκτασης. Σε πολλές χώρες όμως παραμένουν πολλά τα προβλήματα και οι προκλήσεις και σε διάφορους τομείς. Η ανάπτυξη δεν ε, ε, είναι προ όφελο όλων των πολιτών και όλων των κρατών με τον ίδιο τρόπο. Κάποια κράτη-μέλη ακόμα έχουν υψηλή ανεργία και υψηλή φτώχεια. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη το εισόδημα των οικοκυριών παραμένει χαμηλότερα ε, από το επίπεδο του 2008. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και αποκλήσεις στους κοινωνικούς δείκτες και την απασχόληση. Ας πούμε η απασχόληση παραμένει χαμηλή για το ε, τους εργαζομένους που έχουν χαμηλή δίκευση και δεν έχουν γεννηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν και διαφορές στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες επιμένουν. Επίσης, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραμένει πρόβλημα προς επίλυση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες αυτές οι προκλήσεις και άλλα προβλήματα μακροπρόθεσμα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλαγή, ε, την ψηφιοποίηση, την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, την παγκοσμιοποίηση και την κύραση του πληθυσμού, μας καλούν για περαιτέρω δράση για να έχουμε μεγαλύτερη κοινωνική σύγκληση. Επίσης, η μελέτη για την ετήσια ανάπτυξη μιλάει ότι ε, υπάρχουν προβλήματα ε, σε χώρες με ψηλό χρέος, ε, προβλήματα προσαρμογής δηλαδή. Υπάρχουν και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, εντάσεις και υπάρχει και αντίκτυπος του Brexit. Σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως διαπιστώνουμε ότι έχουν επιβραδυνθεί. Η σε αυτή η έκθεση επίση τονίζει ότι είναι σημαντικέ οι εθνικέ μεταρρυθμίσει για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η καταπολέμηση των αποκλεισμών και η θεσμική ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, στόχος αυτής της μελέτης είναι να θέτουμε κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την αντίστασή μας και την αντοχή μας σε μελλοντικού κραδασμούς να καταπολεμούμε τους αποκλεισμούς και καλούμε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τις επενδύσεις, ε, βεβαίως ε, διατηρώντας πάντα τη χρηστή ε, φορολογική και δημοσιονομική πολιτική. Οι επενδύσεις παίζουν ροκλειδί, ε, πρωταγωνιστικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομία. Και επενδύσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με έργα υποδομής, αλλά και κυρίως με τους πολίτες. Η σημερινή συγκυρία επίσης απαιτεί ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και αρχές του να γίνουν πράξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η πολιτική, οικονομική και κοινωνική αντοχή και ανθεκτικότητα κυρίως της Ευρωζώνης. Η πρόταση λοιπόν για την Ευρωζώνη που είναι και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από την αρχή ως μέτρο καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν δράση έτσι ώστε να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις ε, που θα θωρακίσουν την αντίσταση και την αντοχή τους μειώνοντας ε, τις ε, περιφερειακές αποκλήσεις και βοηθώντας τη σύγκληση για να βελτιωθεί η αγορά, να επενδύσουμε σε δεξιότητες και προσόντα και να προστατεύσουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συσφίξει τους θεσμούς, μάλλον να συνδέσει περισσότερο το ευρωπαϊκό εξάμεινο με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ας πούμε, το επόμενο εξάμεινο θα ε, εστιάσουμε στην εκτίμηση ε, των αναγκών για επενδύσεις και ε, έτσι θα καθοδηγήσουμε τα επενδυτικά προγράμματα για την επόμενη περίοδο. οι διάφορες εκθέσεις ε, θα μας βοηθήσουν και θα μας εμπνεύσουν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Και τέλος, θέλω να καλωσορίσω την Ελλάδα ε, στη διαδικασία του εξαμήνου. Έχει ε, επανέλθει πλήρως και τέλη Φεβρουαρίου θα καταρτήσει σχετική έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως για όλα τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Βγήκε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο από τα μνημόνια Και τώρα κάθε τρεις μήνες θα δημοσιεύεται έκθεση με ε, τις εκτιμήσεις. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα ακόμα υποφέρει από την κληρονομιά της κρίσης, αλλά τώρα ε, έχει σταθερή ανάπτυξη, ανακάμπτει αγορά εργασίας και σταδιακά βελτιώνεται η κοινωνική κατάσταση και αυτό φυσικά μας χαροποιεί. Um, Επίσης θα ήθελα να σας πω κάτι ακόμα για την Ελλάδα, γιατί συχνά αυτό κυριαρχούσε στη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης, δείχνουν οι εκθέσεις ότι υπάρχει και αρκετός φορολογικός μάλλον δημοσιονομικός χώρος στην Ελλάδα για να μην χρειάζονται πλέον οι περικοπές των συντάξεων που είχαν προεξοφληθεί και προαποφασιστεί. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί θα είχε και πάλι συνέπεια μια περικοπή των συντάξεων ε, στο εισόδημα ε, των συνταξιούχων που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο και είναι στο κατόφλι της φτώχειας. Υπάρχει λοιπόν αρκετό δημοσιονομικό περιθώριο έτσι ώστε να μην γίνουν οι περικοπές των συντάξεων που είχαν προ και αυτό είναι πάρα πολύ καλά νέα για τον ελληνικό λαό. Η σημερινή οικονομική συγκυρία, πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τι μεταρρυθμίσει και να θέσουν τα θεμέλια για μια ανάπτυξη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμού. Με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και τη κοινωνία των πολιτών. Τη δέουσα συμμετοχή. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν και να χαράξουν τις σωστές πολιτικές, αλλά θα γίνει και κτήματος αυτή η πολιτική και το αποτέλεσμα ε, το κοινωνικό και το οικονομικό θα είναι πολύ καλύτερο. Σε ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσμένω να ακούσω τις απόψεις σας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πολλά θετικά α, ακούμε, πολλά θετικές ειδήσει. Ε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας. Ε. Η Επιτροπή μας προφανώς ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στους συντονιστές. Και μετά μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Ο κύριος Κάζα να πάρει το λόγο από το ΕΛΚΑ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και καλημέρα επίτροπε συνάδελφοι. Και γενικά ναι, συμφωνώ με την εκτίμηση της Επιτρόπου η, η οικονομικοί δείκτες, ε, οι δείκτες ανεργίας στην Ευρώπη είναι πιο φετικοί τώρα, αλλά η οικονομική ανάπτυξη ήδη φαίνεται ότι επιβραδύνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις τώρα, τώρα που οι οικονομικές συνθήκες είναι ακόμα ευνοϊκές. Οι πιο πολλοί δείκτες έχουν επιτέλους ξεπεράσει τα επίπεδα προκρίσης. Παρά όλα αυτά όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καθορίσει μηχανισμούς υποστήριξης για τα κράτη-μέλη για να επιστροφθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό. Να περάσω στο ερώτημα που έχω να κάνω για την πρωτοβουλία για την αλληλεγγύη των νέων και από τι πρόσφατες διαπραγματεύσει για τον προϋπολογισμό. Η πρωτοβουλία αυτή για την ενεργεία των νέων φαίνεται ότι διατηρεί την ισχυρή θέση του και στον 2019 στον προπολογισμό και στο επόμενο και στο πουδουπού. Επιφέρει αποτελέσμα το πρόγραμμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά έχει και ορισμένα προβλήματα, ορισμένε αδυναμίε. Πώ θα ενισχύσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υλοποίηση τη ε, εγγύηση για του νέου, προκειμένου να απορροφείτε να καλύτερα, να καλύτερα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι συχνά δεν θεωρείται αρκετά σκόπιμο και ευνοϊκό να ε, προσλαμβάνονται νέοι. Κυρία Γιονγκέριους από τους Σοσιαλιστές, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία μια και τελειώνει και το έτος και είναι και εδώ η Επίτροπος, να κάνω μια απολογισμό του περασμένου έτους και να ξεκινήσω με ε, τα συγχαρητήριά μου. Γιατί πραγματικά, αν ε, κοιτάξουμε τι έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, θεωρώ ότι έχετε κάνει μεγαλύτερο έργο από την προκατοχή σας και ήταν πολύ ε, καλή συνεργασία στα πλαίσια της οδηγίας για τους αποσπασμένους και για τις ε, ε, Συνθήκε στο συντονισμό σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε μπροστά μα, αλλά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω σε κάθε περίπτωση γιατί πραγματικά καταβάλλετε μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Σήμερα, λοιπόν, με το κείμενο αυτό που έχουμε μπροστά μας, ε, ε, ε, Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο να, αν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας και κατά πόσο να, ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Φυσικά και όχι. Εδώ το θέμα της ισορροπίας ε, επαγγελματικού και προσωπικού βίου δεν είναι αυτονόητο ούτε στη δική μου χώρα και σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες κοιτάνε να δούμε πώς θα τα εξισορροπήσουμε αυτά και προφανώς στην αγορά εργασίας έχει σημασία αν λένε Μαρία ή Φάτιμα δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο ο συνάδελφος ο κ. Κάζα ανέφερε στο θέμα της ανεργίας των νέων πολύ υψηλή σε όλη την Ευρώπη αυτό που διαρωτώ είναι μήπως στο σημερινό κείμενο και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό άλλωστε, μήπως λείπει η αναφορά στις 20 αρχές του Γκέτεμπορκ. Μήπως θα έπρεπε να εργαστούμε πολύ πιο σκληρά για να προωθήσουμε τα σημεία αυτά. Αυτό θα το βάλουμε φυσικά και στο ψήφισμα. Νομίζω ότι θα βοηθούσε αν τα σημεία αυτά του πυλώνα έμπαιναν και στον προϋπολογισμό και στο AGS. Και θα ήθελα λοιπόν αυτό να συνεχίσει να αποτυπώνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Τρεμπέσιος από το ECR. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε σήμερα εδώ να ακούσει και να απαντήσει ερωτήσεις μας παραδοσιακά ήθιστε να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα εδώ και νομίζω ότι παρότι τα προβλήματα που έχουμε στα θέματα μας ε, προηγούνται της κρίσης, αν κοιτάξουμε τα στοιχεία της Ιταλίας και της Ισπανίας, πάλι δεν δίνουν ε, ενθαρρυντικά μηνύματα. Μπορεί να κάνατε μια καλή αξιολόγηση για την κατάσταση στην Ελλάδα. Αν κοιτάξουμε όμως τις συστημικές τράπεζες και τα δεδομένα τους, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τέτοια αισιοδοξία. Το ίδιο και με την ε, Γαλλία διαπιστώνουμε και με τις ε, ε, που τελικά σταματούν ή τουλάχιστον αναστέλλονται εν ώψη των κινητοποιήσεων των κίτρινων ε, γυλαίκων η καινοτομία και όλα αυτά τα θέματα και τα στοιχεία τα σχετικά με την ανάπτυξη βλέπουμε να έχουν καμφθεί αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά αναφέρατε το Brexit. Φοβόμαι πάντως ότι τα στοιχεία του 2016 θα δώσουν πολύ πιο αρνητική εικόνα. Ήδη η BlackRock σήμερα έκανε μια σχετική αναφορά και έκκληση για ανάκληση των ε, ποσών που υπάρχουν στις αγορές ευρώ γιατί θεωρεί ότι είναι κακές οι προοπτικές. Διερωτώ με λοιπόν πόσο ασφαλής είναι η εικόνα για τη Γαλλία, για την Ιταλία και τι έχετε να πείτε για τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Μακρόν προς τα κίτρινα γυλαίκα που μας δείχνουν ότι του χρόνου δεν θα μπορέσει να, για το επόμενο του δηλαδή ο προπολογισμό του δεν θα είναι σύμφωνος με τις ε, δεσμεύσεις του. Επίσης, η πραγματική μισθή πρέπει να είναι ε, σύμφωνη, με, είναι σύμφωνη μάλλον με τις πραγματικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Αν όμως ε, θέλουμε να τους προσαρμόσουμε στην, στην αναπροσαρμογή, την τιμαριθμική, τότε θα αυξηθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και διερωτώ με τι σκοπεύετε να κάνετε για να διαφυλάξετε την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωζώνη και να τη βελτιώσετε μακροπρόθεσμα. Η ενέργεια των νέων αναφέρθηκε. Τι μέτρα σκοπεύετε να εισαγάγετε για να κάμψετε μακροπρόθεσμα την ανεργία των νέων. Και ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας. Κύριος ε, Κάλλιες Τσάμπον. Άλντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλημέρα σας. Και πάλι καθώς τελειώνει η βουλευτική περίοδος με μεγάλη χαρά και ε, τιμή σας βλέπω εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερως για τις τοποθετήσεις σας. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ θετικό και δεν θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου γλώσσα του Θερβάντες για να σας ε, απευθύνω το λόγο στα γαλλικά ώστε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία. Είμαι λοιπόν ε, ιδιαίτερα ικανοποιημένο για λογαριασμό όλων μας ως προς την απαόφαση που ελήφθη όπως άλλωστε επισημαίνετε και εσείς, ότι η οικονομία και, η και τα κοινωνικά μελήματα πρέπει να προχωρούν όταν κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα χέρι με χέρι. Διότι δεν υπάρχει κοινωνικός αντίκτυπος που να μην σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση και τούμπαλιν. Έτσι λοιπόν ε, ένα οικονομικό, κοινωνικό μια, κοινωνική οικονομική σύνοδος ε, κορυφής έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με την εισαγωγή του scoreboard μετατρέπεται την κοινωνική σύνοδο σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και το καταφέρατε πολύ καλά αυτό. Κάτι ακόμη και Εδώ και 4,5 χρόνια αυτά τα πράγματα τα υποστηρίζω εγώ, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε και καθώς δεν έχω τόσο χρόνο θα περιοριστώ στο εξής, ότι ίσως παρέσασταν ε, ε, ευνοϊκοί σε ορισμένα, όχι τόσο βέβαια στην, τρί, στην τρίμηνη έκθεση για την Ισπανία, αλλά ίσως παρέσετε επίοικης σε ένα σημείο που έχει τεράστια σημασία και θα το βρούμε μπροστά μας. Συμφωνώ στα όσα είπατε με την ανεργία, και η πατρίδα μου έχει 15%, εντάξει μπορεί να έχουμε και να εξελίσσεται, άρα πάση έχουμε 13 δείκτε κτλ. Αλλά, αλλά παραμένουν οι ανισότητες και ενισχύονται και από εκεί προέρχεται και η δυσφορία και ε, τα προβλήματα τα κοινωνικά που μπορούν να αποβούν, εις, ε, να αποβούν επιζήμια τελικά για τις δημοκρατίες μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και είναι προφανές ταυτόχρονα αν κοιτάξουμε δηλαδή τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και τώρα σας μιλώ όχι στους Ισπανούς αλλά ως Ευρωπαίους. Αν δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό που ονομάζεται κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στην Ευρώπη, είναι μια αντίδραση απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αρέσει στον πολίτη μας. Λέει ο κ. Μακρόν ότι εντάξει βρισκόμαστε σε μια αποκατάσταση, αναδιάταξη οικονομική, κοινωνική, κοινωνικο-οικονομική, έστω. δεν νομίζω ότι μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αντίστοιχα σε άλλες χώρες από την Ισπανία μέχρι τη Βουλγαρία. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια τεράστια δυσφορία. Έχουμε να κάνουμε με πολλές θυσίες που στον πολίτη με ε, διατήρηση όμως των αδικιών, αδικιών που έχουν διωγγωθεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση και άρα για να ολοκληρωθεί και να τελειωθεί αυτή η, να ολοκληρωθεί αυτή η καταπληκτική δουλειά που λέγατε ότι είναι κάναμε σημαντικά πράγματα αλλά δεν αρκούνε. Μα νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερα να απευθύνουμε, ε, να, κρούσουμε τον κόδωνα κινδύνου στα όσα συμβαίνουν και στα κράτη-μέλη και στα όσα διαπιστώνει. Το τελικά έχουμε δείκτες ε, καλούς οποίοι όμως διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα κράτη έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι σε κάποια άλλη. Άλλα και έτσι μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα τα νούμερα και κάποιοι να γίνονται πιο πλούσιοι, αλλά οι αδικίες, οι κοινωνικές, οι ανισότητες, οι κοινωνικές ε, είναι πολύ, είναι πολύ υψηλές σε πολλές περιπτώσεις και πολύ σωστά αναφέρεται και την διάσταση της φορολογίας γιατί η ανισότητα δεν θα αντιμετωπιστεί με ένα φιλοδόρημα ή με την ε, χορήγηση επιδομάτων ή άλλων κονδυλίων πρέπει να αντιμετωπιστεί φορολογική αδικία. Και πρέπει εκεί να δώσουμε έμφαση, γιατί αυτό είναι το ευρωπαϊκό πνεύμα, να καταλάβει ο πολιτή ότι όταν δουλεύει, δουλεύει όχι για να γίνει κανείς πιο πλούσιος, αλλά για να εξασφαλίσει μια κοινωνία πιο ισότιμη και πιο δίκαιη. Ευχαριστώ πολύ. Η Γκουέ δεν βλέπω να έχει εκπροσώπηση εδώ, κάνω λάθος. Τζιν Λάμπερτ, πράσινη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Και θα, το συνδυάσω θα τα συνδυάσω με αυτά που είπε και η επίτροπο στη γύρανση δηλαδή, που συναφής είναι και με την ανεργία των νέων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτούς που παρά είναι γέροι, ώστε, να τους καλύψει η, ώστε δεν τους καλύψει τελικά η πρωτοβουλία για τους νέους, αλλά που πάλι δεν είχαν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουν ε, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και άρα και μάλιστα ποτέ δεν είχαν μια απασχόληση που να ανταποκρίνεται και να ανακλά τις δεξιότητές τους, δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν ποτέ από μόνιμη απασχόληση. Για αυτούς τι κάνουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ε, στεγανά που να αποκλείουν κάποιον ο οποίος έχει χάσει μια ευκαιρία σε ένα γύρο της ζωής του ε, από την ε, απόλαυση δυνατοτήτων σε κάποια άλλη φάση. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια των ε, ενηλίκων που έχουμε παραδείγματι που δεν έχουν ούτε, τα, ούτε τις γνώσεις γραμματικές, αριθμητικές ή ψηφιακές που θα τους επέτρεπαν να προχωρήσουν σε μια επόμενη φάση μέσα στην ψηφιακή αγορά και άρα πολλές είναι οι δυσκολίες που μπορούμε να διαπιστώσουμε για αυτές τις κατηγορίες των πολιτών σε όλα τα σε πολλά κράτη-μέλη. Επίσης αναφερθήκατε στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής Και βεβαίω υπάρχει εκεί μεγάλο δυναμικό, αναφέρεται και από διάφορε εκθέσει, κυκλική οικονομία κτλ. Πιστεύετε ότι οι σχετικέ δεξιότητε, οι δεξιότητε που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία, ε, παρακολουθούν το δυναμικό επέκταση των δυνατοτήτων ε, της ε, δραστηριοποίησης στον χώρο της κλιματικής αλλαγής ή έχουμε χάσει το τρένο. Άλλο επίσης, ανισότητα, λέξη που επισήμεναν πολλοί συνάδελφοι. Πρώτον, στη στέγη. Η στέγη ε, προσλαμβάνει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις με ένα κρατημέλι. Εάν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει το τίμημα, ε, το αντίτιμο μάλλον μιας στέγης αξιοπρεπούς, μια στέγης ευχάριστης, αυτό θα έχει συνέπειες σε πολλά άλλα κοινωνικά θέματα, βέβαια και στην ανάπτυξη των ίδιων των παιδιών. Έτσι λοιπόν διαρωτώ με, δίνουμε αρκετή έμφαση στο στόχο της ανάπτυξης, στο κομμάτι της ε, στέγης. Κυρία Άουγκια, η ευθύτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της βουλευτική περίοδου και πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη χαρά από ήμουν μέλος της Επιτροπής. Ε, Απασχολήσω όχι μόνο γιατί είχα την ευκαιρία να δω σε συνεργασία με τους συναδέλφους ότι μπορούμε να δείξουμε τη βούληση να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών αλλά και γιατί στο πρόσωπό σας αναγνωρίζω φιλοδοξία που δεν έχω δει να εκδηλώνουν άλλοι επίτροποι. Δουλέψαμε λοιπόν όχι μόνο με φιλοδοξία, αλλά και με ζήλο, με δυναμικό, με ικανότητα, με στρατηγικό όραμα σε σημαντικές, πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις. Ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για το, η προστασία των εργαζομένων, την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες. Και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο να πούμε ότι πρόκειται για μια επιτροπή απασχόλησης. Εδώ η επιτροπή που εμείς ε, ε, συνθέτουμε, είναι κάτι περισσότερο και μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και με άλλες εκθέσεις βεβαίως, συμφιλίωση επαγγελματικού και οικονομικού βίου που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη με την γύρανση του πληθυσμού χρειάζεται συγκεκριμένε απαντήσεις, χρειάζεται την υποστήριξη με τη φροντίδα προς τις οικογένειες, προς τα άτομα. Ε, χωρίς να υποστηρίζω όλες τις προτάσεις πάντα βλέπω ότι υπάρχει φιλοδοξία. Το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας μοιραζόμαστε και έχουμε στόχους που μπορούμε να ε, επιτύχουμε με τις τεράστιες βέβαια και ανισότητες που έχουμε ανάμεσα στους πιο φτωχούς και τους πιο πλούσιους. Ε, τη δική μας την πρόταση για ένα εισόδημα το πολίτη που ξέρω ότι υποστηρίζετε εσείς γιατί είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί το φάσμα της ανεργίας και της φτώχειας. Πρόκειται για ένα επίδομα λοιπόν, για μια λύση που μπορούμε να θέσουμε σαν στόχο σε μια χρονική στιγμή όπου κάποια δειλά μόνο βήματα διαπιστώνουμε ακόμα προς την ανάκαμψη, ενώ είναι πολύ φτωχοί, υπερβολικά πολύ οι που χρειάζονται άμεση υποστήριξη. Ταυτόχρονα χρειάζεται και μεταρρύθμιση του συστήματος ταξιοδότησης ώστε να διαφυλαχθεί μια ομαλή μετάβαση ε, και παράδοση της κοιτάλης των γενναίων που θα προστατέψει τους πιο ηλικιωμένους αλλά και θα επιτρέψει ταυτόχρονα στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι η ελπίδα, η αισιοδοξία που από κοινού μοιραζόμαστε μια δουλειά σταθερή, συνεπής, μια δουλειά θαραλέα που αναπτύσσουμε από κοινού μπορεί να μας οδηγεί στους στόχους. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μπορεί μερικές φορές να μας απαγοητεύει ο κόσμος όπως ε, πηγαίνει, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή μας έδειξε ότι μπορεί κανείς με θάρρος και παρησία να κάνει δουλειά αποτελεσματική για τον πολίτη και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και επιτρέψτε μου μια αναφορά στην Ελλάδα Μερικές φορές αναφέρεται ότι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, τα μνημόνια, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, ήταν απαραίτητα ε, μέτρα, μέτρα ουσιαστικά αναπόφευκτα. Αλλά θα ήθελα από την Επιτροπή μας να απευθύνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα κατέστη πειραματόζω, έγινε ένα πείραμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα, μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα για τους πολίτες μας και για τα κράτη μας, για τη σύγκληση, για τους θετικούς στόχους που μπορούμε να επιτύχουμε, που μπορούμε να επιτύχουμε όμως ε, με διαφορετικές μεθόδους. Αν λάβουμε υπόψη, όπως είπατε και εσείς, ότι πριν να γίνονται οι μεταρρυθμίσεις πρέπει πάντα να αξιολογείται η συνέπεια, το σύνολο των συνεπειών τους. Ευχαριστώ. Ενφ δεν βλέπω εδώ. Κυρία Μαγάν Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι σας εκδιάζουν για την εργασία σας. Πρέπει να πω ότι μας κάνετε περήφανους που εργαζόμαστε εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Από τότε που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ΕΜΠΕΛ θεωρεί το μα, υποδιαδέστερη άλλων επιτροπών. Από τη δική σας όμως εργασία, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας κινητοποιηθήκαμε για να κερδίζουμε ψηφοφορίες και να προωθούμε τις ιδέες μας, καταφέραμε να κατακτούμε πλειοψηφίες στην Ολομέλεια προς την κατεύθυνσή μας, πράγμα που δεν ήταν καθόλου βέβαιο. Ήσασταν λοιπόν ένας κινητήρας, μια κινητήρια δύναμη για την ε, κοινωνική Ευρώπη και μας βοηθήσατε να προχωρήσουμε πάρα πολύ και όλοι μαζί προωθήσαμε την ιδέα μιας κοινωνικής Ευρώπης στα μάτια των συναδέλφων μας στην Ολομέλεια. Και πραγματικά γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Γιατί όταν έχεις κάνει τέτοιο μεγάλο βήμα θα πρέπει να ε, τηρήσεις τις θέσεις αυτές και να συνεχίσεις προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να, να, να αναφέρω, συγγνώμη, και το είπε και η συνάδελφος Τζιν Λάμπερτ, επιγραμματικά είναι το θέμα ε, του μέλλοντος, οι δεξιότητες και τα προσόντα. Ε, μας παρουσιάζεται σημαντικά στοιχεία για τους δείκτες, η κατάσταση βελτιώνεται για την απασχόληση κτλ. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε ότι τα επόμενα έτη θα ε, εμφανιστούν νέα επαγγελματά, νέες ε, δεξιότητες θα γίνουν απαραίτητες. Και αυτή η κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει να αλλάξει τελείως τον τρόπο κατάρτισης και το μοντέλο το ίδιο κατάρτισης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις. Και αυτό εμείς θα πρέπει να το πλαισιώσουμε και να το υποστηρίξουμε, αλλιώς θα ξαναπέσουμε στην παλιά προβληματική κατάσταση. Για να σταθεροποιηθεί λοιπόν αυτή η εικόνα που μας έχετε σκιαγραφίσει, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου τις δυνάμεις μας για να προετοιμάσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας dans le milieu ε, ε, ε, Με αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και μη επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, το τονίζω αυτό, για να ξεφύγουμε από τα στάνταρ, διπλώματα, πτυχία κάθε της εκπαίδευσης και να περάσουμε σε μια πιο εγκάρσια, οριζόντια εκπαίδευση για να μην έχουμε νέους ανέργους που θα βρεθούν σε αυτή την απόγνωση. Μας απομένουν λίγοι μήνες ε, συνεργασίας. Εγώ είμαι αισιόδοξη για να δώσουμε και τέτοιες πρόπτικες στους νέους μας. Ζητώ συγγνώμη που θα αποχωρήσω γιατί θα πρέπει να πάω να ευχαριστήσω ε, τους οδηγούς μας και το προσωπικό της εστίασης που εργάστηκαν όλη τη νύχτα μετά την τρομοκρατική επίθεση. Θα συνεχίσω λοιπόν στην πράξη αυτό που κάνουμε εμείς στην Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη κυρία Επιτροπέ και κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, yeah, thank you. You know, um, we have Σας ευχαριστώ και οπότε ξέρετε έχουμε και ένα τέσσερα θέμα στην ημερική διάταξη. Δεν θα προλάβουμε αν ε, μιλάτε παραπάνω από 1,5 λεπτό. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά προσπαθείτε να μην επαναλάβετε αυτά που έχουμε ήδη ακούσει. Κυρία Ροντρίγκε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ε, έχω φωνή, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω. Να σας πω τι εννοώ. Εγώ με τους συναδέλφους μου συμφωνώ συμφωνώ όταν υπογραμμίζουν τη σημασία να υπάρξουν αποτελέσματα στην κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά είμαστε ευγνώμονε. Είμαστε ευγνώμονε για το ρόλο που έχετε. Ήταν πραγματικά πολύ καρποφόρα αυτή η πολιτική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να υποβάλω και εγώ το δικό μου ερώτημα. Συζητάμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο με τέτοιο τρόπο προκειμένου να καταστεί μια δυναμική διαδικασία καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων και μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην οικονομική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κεντρικό για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η απάντηση είναι η εξή θεωρώ. Καταρχάς, θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία πολιτικής του εξαμήνου. Τις εκθέσεις αναχώρα, το scoreboard, τον πίνακα με τα αποτελέσματα, τις ε, συστάσεις αναχώρα. Με ισχυρή επικέντρωση στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και εδώ πιστεύω ότι οι επενδύσεις, ε, μάλλον η αξιολόγηση επενδύσεων αποτελεί καλό εργαλείο. Δεύτερο σκέλος στην απάντηση χρησιμοποιώντας τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα για την καταπολέμηση των ε, οικονομικών ανισοτήτων. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων και θα ήθελα να τονίσω ότι αύριο οι Πρωθυπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν στα πλαίσια της Συνοδού τις δυνατότητες οικονομικής ε, ικανότητας της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτή η ικανότητα κοινωνικών επενδύσεων. Αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε. Τελευταίο σημείο. Για το ρόλο της φορολογικής πολιτικής. Γιατί όσο πιο πολύ το κοιτάμε το θέμα, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ότι το τμήμα της λύσης είναι η πιο δίκαιη φορολογική πολιτική και πόρη φορολόγησης ε, για τη χρηματοδότηση των συστημάτων μας στο μέλλον. Αυτά ήταν τα όσα είχα να πω για την επόμενη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέγει η Πρόεδρο, και θα δώσω τώρα το λόγο στην Άκνια Σκακοσλόφσκα Ράντοβιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την Επίτροπο για τι αισιόδοξε αυτέ πληροφορίε που μα δώσατε για τη βελτιωνόμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι γεγονό ότι έχουμε χώρε οι οποίε αναπτύσσονται ταχύτερα στην Ευρώπη και η Πολωνία είναι μία από αυτέ. Φέτο είχαμε 5%, πάνω από 5% οικονομική ανάπτυξη του χρόνου προβλέπεται πάνω από 4%. Είναι ψηλά τα ποσοστά αυτά. Ωστόσο, συμφωνώ ότι δεν είναι τελικά μόνο ο ρυθμός, ε, το ποσοστό ανάπτυξης που έχει σημασία. Θα πρέπει να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη αυτή και ισορροπημένη να φέρνει πραγματική βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, μοντέρνες ιδέες για την ε, πρόοδο χωρίς την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπό γιατί στην έκθεση της δεν τονίζεται τόσο η διάσταση του φύλου. Γιατί όταν μιλάμε για αύξηση της ε, απασχόλησης, ξέρουμε ότι οι υποεκπροσωπούμενες ε, ομάδες στην αγορά εργασίας είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο δραμικό ανάπτυξης. Γιατί εκεί οι ομάδες αυτές μπορούν να συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη και αυτός περιλαμβάνει όχι αποκλειστικά, αλλά βασικά τις γυναίκες, άτομα με ικανότητες, προσόντα, δεξιότητες που μπορούν να συμβάλλουν στην αγορά εργασία. Επίσης, δεν αναφέρεται τίποτα, δεν, δεν αναφέρεται πολλά για το μης ελλημάτων, όπως είναι το ICT, οι μεταφορές. Μιλάμε βέβαια για την ενέργεια, αλλά έχουμε και το μης όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι λείπουν λοιπόν, και δεν προσελκύουν κόσμο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα με νόμιμη μετανάστευση, με προσπάθεια ίσως ε, πρόσληψης ε, από ομάδες υποεκπροσωπούμενες, όπως οι γυναίκες στον τομέα των IT, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι τέτοιες πολιτικές θα βοηθούσαν. Και τέλος, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα της ε, εκπαίδευσης και της κινητικότητας. Όταν μιλάμε για έλλειψη εργατικού δυναμικού από τη μία και ανεργία από την άλλη, μιλάμε για προβληματική ισοκατανομή και αυτό θα ήταν μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει την αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ριμπέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο η Ευρώπη σήμερα έχει καταστεί πιο κοινωνική και όλες αυτές τις υποχρεώσεις ε, Έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή στην Επιτροπή μας και χαίρομαι που μπορούμε να συμβάλλουμε στην ε, πιο δημοκρατική και κοινωνική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετείχα και στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τίθεται το θέμα των ε, κοινωνικών δικτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το πετύχαμε αυτό να μπουν οι δείκτες αυτοί. Και τώρα κοιτάμε λοιπόν πώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή κατά των μακροοικονομικών αποκλήσεων. Και όταν μιλάω για μακροοικονομικές αποκλήσεις, δεν εννοώ μέτρα τιμωρητικά για τα κράτη-μέλη. Όχι. Πολύ πιο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να έχουν την υποχρέωση να καταπολεμούν αυτές τις ανισότητες. Αυτό είναι μια πρόκληση την οποία θα την αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις δικασίες αυτές, θα πρέπει όλα αυτά να συμβαίνουν παράλληλα με τους μικροοικονομικούς παράγοντες. Αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε ανάλυση της ε, κοινωνικής κατάστασης ε, των ε, πολιτών, κατά πόσον, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια κατοικία. Είναι σημαντικό να υπάρχει θετική εντύπωση για τους πολίτες για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν μπορούμε να, θεω... να επιτρέψουμε να θεωρείται τιμωρία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όχι. Ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται μια σωστή τοποθέτηση, μια σωστή αντιμετώπιση. Υπάρχουν δυσκολίες ό,τι αφορά την υλοποίηση σε κάποια κρατημέλη. Υπάρχουν κρατημέλη όπου υπάρχουν ε, πολιτικές και διοικητικέ διαφορές. Υπάρχουν πολλές ε, περιφερειές και περιοχές που είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες διοικητικά και αυτές άμεσα θα πρέπει να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό ισχύει και για τις εξόχως αποκεντρωμένες περιοχές, μια ζώνη από την οποία και εγώ προέρχομαι και έχουν δυνατότητα λοιπόν να συμμετέχουν πολύ πιο δραστικά και ενεργητικά στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σύμβαση για το πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ήδη δυνατότητες ενισχυμένη συμμετοχή των περιφερειών, των εξόχους απόκεντρων περιοχών στη διαδικασία αυτή προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν άμεσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να, να εξισορροπήσουμε τα θέματα αυτά, προκειμένου να συμμετέχουν όλε οι περιοχέ. Κυρία το πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σα ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ηγηθήκατε των εργασιών μα όλο αυτόν τον χρόνο σήμερα που είναι η τελευταία μας ε, συνεδρίαση και εσάς κύριε Επίτροπε. Να σας ευχαριστήσω διότι στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο να σας ευχαριστήσω διότι στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο αντιλήφθημε πόσο σημαντική είναι η κοινωνική Ευρώπη. Έγινε αντιληπτό η σημασία της κοινωνικής Ευρώπης, προχώρησε ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίησή του. 18 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στο όριο της φτώχειας. Συζητούμε τα, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ψηφίζουμε εμείς ένα νέο μέτρο που είναι εγγύηση για τα παιδιά, ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, για την οποία θέλουμε να προβλέψουμε κονδύλια 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ και θα ήθελα να ξέρω αν εσείς ως Επίτροπος, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει την ε, ευρωπαϊκή αυτή εγγύηση για τα παιδιά για να καταπολεμήσει τη φτώχεια των, παιδιών. Λέτε μάλιστα ότι κινδυνεύουν περισσότερο από αποκλεισμό τα παιδιά που έχουν αναπηρία σε σχέση με αυτά που έρχονται από τις υπόλοιπε κοινωνικές ομάδες. Οι περιφερειακές ανισότητες επίσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αναφέρατε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση κατάστασης, αλλά η κατάσταση πραγματικά βλέπετε ότι αλλάζει στα κράτη-μέλη. Βλέπετε κάποιες εξελίξεις όταν έχουμε όταν βλέπετε ότι έχουμε διαφορές στις ε, συντάξεις τόσο μεγάλες μέχρι και στο διπλάσιο. Κυρία Λόπε Φόντανιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ε, και εγώ προσωπικά πρέπει να σας πω ότι είναι η δεύτερη θητεία μου και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ε, ότι υπήρχαν ε, θετικές εξελίξεις ε, για τα κοινωνικά και τα εργασιακά ζητήματα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και είμαι πεπισμένη ότι είχε πολύ μεγάλη σχέση η ίδια Επίτροπος με αυτή την ε, κυριαρχία και την προβολή την καλύτερη των κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων. Γίνανε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φυσικά βελτίωσαν ε, γενικώ ε, στη βελτίωση της ευημερία και των εργασιακών συνθήκων. Βεβαίως έχει ακόμα μείνει πολλή δουλειά ε, για την ανεργία και κυρίως την ανεργία των νέων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Και συμφωνώ ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, προβλέπεται σχετική δράση και σχετικό σχέδιο μάλιστα. Εμένα όμως με ανησυχεί κάτι άλλο. φαίνεται ότι βρισκόμαστε λίγο στα όρια της ανάπτυξης. Έχει εξαντληθεί και μπορεί να επιδεινωθεί η ε, οικονομία τα επόμενα έτη. Και γνωρίζουμε ότι αν επιδεινώνεται και όταν επιδεινώνεται η οικονομία, δυστυχώς επιδεινώνονται και οι κοινωνικές πολιτικές. Έρχομαι λοιπόν στην ερώτησή μου σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Και καλά κάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τα κοινωνικά και τα εργασιακά ζητήματα. Και δεν θα πρέπει αυτά να ε, είναι ε, λιγότερο σημαντικά από τα οικονομικά θέματα. Θα πρέπει και στο μέλλον να μην χαλαρώσει αυτή η προσοχή. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στην Πρόεδρο συμφωνώ ότι έκανε θαυμάσια δουλειά ε, σε αυτή τη τετραετία που προείδρευε και ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Τόμας Μαν. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ήθιστε οι ευρωβουλευτές να επενούν και να εγκομιάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα αυτό είναι διαφορετικό. Αγαπητή Μαριάνε, ε, συγχαρητήρια. Έτσι και όσοι είσαι πρώην Ευρωβουλευτής. Είσαι πάντα παρούσα, ε, με δημιουργικότητα, πολύ εργατική. Και αυτά πρέπει να τα λέμε, όχι επειδή είμαστε τόσο καλοί και συμπαθείς, αλλά γιατί περιγράφουμε και αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Και αυτό <laughs> βεβαίως σε χαροποιεί και σένα, σε επίτροπο. Ε, βοηθήσαμε τους νέους και η δουλειά μας ακριβώς είναι να βοηθούμε τους νέους, εγγύηση για την νεολαία. Ε, είναι ε, εμπορικά σήματα, ε, πραγματικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αγαπητή Μαριάννα, έχουμε και προβλήματα με την ανεργία τη μακρόχρονη ανεργία, γιατί ακούμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε λόγο, έχουμε λίγες ε, προσφορέ, ε, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην αγορά εργασία. Αυτά μα λένε οι άνεργοι. Ε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη απάντηση. Μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα δοθεί αυτή. Και δεν είναι μόνο χρηματικό το θέμα, αλλά θα πρέπει να του ενθαρρύνουμε αυτού του μακροχρόνιου ανέργου, να του λέμε ότι δεν του έχουμε αφήσει στη μοίρα του, δεν του έχουμε καταλήψει. Αυτό με απασχολεί. Εγώ είμαι σκιώδη ηγητή για την ε, έκθεση για το Erasmus Συν και αυτό είναι ε, ε, ένα καταπληκτικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε μόνο ε, τους φοιτητές αλλά και τους μαθητευόμενους από τις εταιρείε που να μπορούν να κυκλοφορούν, να συλλέγουν, να αποκομίζουν επαγγελματική εμπειρία και να μιλάμε καλά, η επαγγελματική κατάρτιση τώρα είναι κάτι δευτερεύον. Στο Εράσμος ΣΥΝ ελπίζω να συμφωνήσουμε και με άλλα όργανα και αν γίνει αυτό έχουμε προχωρήσει ακόμα ένα βήμα. Μπράβο Μαριάννα. Πολύ καλή δουλειά. Ακούς τους επένους. Και πραγματικά πολύ ε, θα προσεύχονται για σένα. Ο κύριος Ροσφόρ, ε, θα είμαι ε, σύντομος και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά να πω κάποια ε, συμπληρωματικά πράγματα. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε, αλλά γιατί σας συγχαίρομαι. Δεν συγχαίρουμε εσάς προσωπικά, αλλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Γιούνκερ, που κατάλαβε ότι τούτη εδώ η Επιτροπή στο δεύτερο ημισή της θητείας θα έπρεπε να δώσει μια διαφορετική εικόνα για την πολιτική και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι έδωσαν οι προηγούμενες επιτροπές και εσείς προσωπικά αλλά και με άλλους επιτρόπους και άλλες γυναίκες επιτρόπους με την κυρία Βεστάγκερ ας πούμε είστε από τις γυναίκες επιτρόπους ε, που, ε, που είστε πραγματικά το καμάρι μας και το λέω πέρα από το προσωπικό μήνυμα είναι και πολιτικό το μήνυμα αλλά έχουμε και πρόβλημα στη συνέχεια να πείθουμε τους πολίτες. Το γνωρίζετε κι εσείς ότι προχώρησε η κοινωνική Ευρώπη. Και δυστυχώς ως Γάλλος με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες ομολογώ ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβάλλουμε και να τονίσουμε τις πρόοδους της κοινωνικής Ευρώπης. Και τα θέματα που σήμερα έχουν τελειώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ολομέλειας θα πρέπει να ε, ε, εκτελεστούν εγκαίρως, ας πούμε, η εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι για τις λεπτομέρειες, αλλά να προωθηθεί αυτό το θέμα και να το καταλάβουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι, γιατί έρχονται και εκλογέ, ότι έχουμε προχωρήσει, έχουμε κατακτήσεις πετύχει και συχνά ομολογώ και δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών με βαριά καρδιά ομολογούν και αυτοί ότι προχωρεί η Ευρώπη και όχι ήδη. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω και απαντώ κάπως σε μία συνάδελφο και θέλω να σας κάνω και μία πρόταση αυτό. Η μεγαλύτερη απειλή σήμερα για τα κοινωνικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ότι θα ξεφύγει λίγο η Γαλλία στις δαπάνες σε σχέση με τον προγραμματισμό της. Πρώτον, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να μελετήσει ε, τον ε, γαλλικό προπολογισμό. Δηλαδή, δεν αρκεί ένα χρόνο να ξεφύγει λίγο παραπάνω από το 3% για να δημιουργηθεί κρίση. Χρειάζεται και δεύτερο οικονομικό έτος. Και ελπίζω να μην ξεπεράσουμε το δεύτερο αυτό κατόφλι που είναι 3,5% του ελλείμματος του χρόνου. Να μην λέμε λοιπόν ότι αυτό το βασικό πρόβλημα, το σημαντικότερο πρόβλημα για τα κοινωνικά στην Ευρώπη είναι οι συνέπειες από την άνοδο του λαϊκισμού σε διάφορα κράτη-μέλη, από την άνοδο του προστατευτισμού παγκοσμίω. Εγώ εδώ θέλω να πω και να διατρανώσω ότι και τα δύο αυτά, και ο προστατευτισμός και ο λαϊκισμός, συγγνώμη να τελειώσω, ε, ε, ε, μας δείχνουν καθημερινά μελέτες ότι το Brexit ποιος το ψήφισε και ποιος απειλείται περισσότερο αυτοί που έχουν κοινωνικές ε, δυναμίες. Άρα δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά προβλήματα που κυριαρχούν και είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες για τα κοινωνικά. Ζητώ συγγνώμη Πρόεδρε. Ναι ξέρετε όμως κλέβετε λεπτά από το επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και παρακαλώ την κυρία Ρενάρα αυτό το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς τη Μαριάν, όπως και άλλοι συναδελφοί, για τη δουλειά της στην Επιτροπή. Δεν ήταν καθόλου απλά τα πράγματα. Κάποιοι επίτροποι οπωσδήποτε δεν συμμερίζονται τις θέσεις της ως προς τους κοινωνικούς δείκτες και τη χρήση του στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κύριε Επίτροπε, το είπατε κι εσείς, δεν είναι το άπαν η ανάπτυξη υπάρχουν ανισότητες, ανισότητες οι οποίες ε, στηρίζονται στις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο στις περιφέρειες και μάλιστα σε ορισμένες χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία μεγάλη οικονομική δύναμη στην, ε, στην Ευρώπη ε, γνωρίζει πολύ σημαντικές ακόμη ανισότητες οικονομικές και κοινωνικές και ανάπτυξης και βεβαίως και, στον τομέα, και στην τομεακή διάσταση διαπιστώνονται σε τομεακή ανάγνωση διαβάζονται ακόμα πολλές ανισότητες. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι κλάδοι της οικονομίας που μπορεί να είναι πιο πρόσφοροι για το μέλλον, που μπορούν να στηριχθούν καλύτερα για το μέλλον ή ποιοι είναι εκείνοι που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στο μέλλον. Πολλές φορές μιλούμε για τη στήριξη και τη μετώπιση των ανισοτήτων με βάση την προσέγγιση στο πρόσωπο, στο άτομο, αλλά νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε και διάφορους τομείς ή κλάδους οικονομίας. Είπατε ότι η απασχόληση έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ πιο μεγάλη όμως η ποιότητα στην εργασία έχει σημασία. Έτσι λοιπόν εάν έχουμε όλο θέσεις εργασίας μηδενικών ορών, ορισμένου χρόνου, μερικού χρόνου, αυτό οδηγεί σε φτωχοποίηση του πολίτη και σε αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερω. Η αύξηση των ενισχύσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία με το σχέδιο Juncker, επί παραδείγματι, που όμω ενισχύει τι πιο ισχυρέ οικονομίε, ενώ για τι πιο αδύναμες δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη και σε αυτό χρειάζονται διορθώσει. Είναι σημαντικοί οι δείκτες λοιπόν και πρέπει να τους αναλύουμε ή να γίνεται η ανάλυση τους σε πολύ πιο ε, λεπτομερή βαθμό για να τους χρησιμοποιούμε καλύτερα. Αλλά θα ήθελα να δω και τι θα κάνουμε με τους δείκτες αυτούς. Πώς δηλαδή αλλάζουμε πολιτική μέσα στο, την πολιτική του εξαμήνου. Και παίρνω δύο χώρες με τα δελτία τους, τη Γαλλία, την αξιολόγηση της το 2017 σχέση με τις βελτιώσεις που παρουσιάζει και τι μας λέει εδώ για, την Επιτροπή, για τη Γαλλία η Επιτροπή και τις βελτιώσεις. Μας λέει ότι ε, είναι ικανοποιημένη για την ενίσχυση της ευελιξίας ε, στην, και την εισαγωγή αυτής στις επιχειρήσεις που επιτρέπουν, όπου επιτρέπεται πλέον οι απόλυσεις, μαζικές απολύσεις, έχουν διευκολυνθεί οι απολύσεις και έχει ελαφρυνθεί η φορολογία των επιχειρήσεων. Δύο από τα πράγματα που αμφισβητούν και καταδικάζουν αυτή τη στιγμή ε, τα κίτρινα κυλέκα. Δύο πράγματα που δεν είναι διατεθειμένοι οι εργαζόμενοι να δεχθούν, δηλαδή την ελάφρυνση τη φορολογία για το κεφάλαιο ε, και την επιβάρυνση φορολογία ταυτόχρονα για τον εργαζόμενο. Την ευελιξία που ε, καλείται να εκδηλώσει μόνο ο εργαζόμενος αλλά ποτέ η επιχείρηση. Και άρα χρειάζεται συνοχή ανάμεσα σε αυτά που λέμε για του κοινωνικού δείκτε και στα όσα κάνουμε όταν προάγουμε κάποιες πολιτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ, Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα είμαι σύντομη, μια και έχω τη δυνατότητα να μιλήσω αργότερα. Ε, θα ήθελα ωστόσο να ε, σύγχαρω την Επιτροπό, να την ευχαριστήσω για την καλή της ε, δουλειά τρεις ε, περιόδους είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Με τη δεύτερη πρέπει να πω ότι είχα χάσει κάθε ελπίδα να δω να προκύπτει από το Κοινοβούλιο η αδίποτε κοινωνική ισότητα και ισοτιμία στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τότε που είχαμε την Λισαβόνα τότε που με το δημοψήφισμα είχαμε υποσχεθεί στους Ιρλανδούς ε, την σημασία που θα έφερνε στις ζωές τους, που θα είχε για τις ζωές τους η εφαρμογή του άρθρου 9 και στην επόμενη θητεία που δεν είχαμε καν τη δυνατότητα να, να επακαλυστούμε το άρθρο 9. Με τα βίας γινόταν μια σε υποσημείωση η παραπομπή. Ωστόσο βλέπω ότι οι δικές σας οι προτάσεις μας επέτρεψαν με την μεγάλη ε, αποτελεσματικότητά τους να φέρουν σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο στη ζωή των πολιτών και τελικά αυτό νομίζω ότι είναι και το νόημα της παρουσίας όλων μας εδώ στη δουλειά αυτή που κάνουμε και γι' αυτό ευχαριστώ και εσάς αλλά και την, Επίτρο, και την ε, Πρόεδρο η οποία καθοδηγώντας τι εργασίες μας μας επιτρέπει να εκδηλώσουμε και να εκφράσουμε με τρόπο απτό τις φιλοδοξίες, ε, τις προσδοκίες μας και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την εννοούμε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε βέβαια που χρειάζεται κάποιες φορές να σταματώ αυτή την τόσο σημαντική, ε, μια τόσο σημαντική παρέμβαση γιατί έχουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Αλλά και εσείς προσπαθήσατε να είστε σύντομοι. Κύριε Τέσσερ, νομίζω ότι 10 λεπτάκια τα έχετε για να απαντήσετε. Αν όχι σε όλες τις ερωτήσεις, πάντως να δώσετε μια αντίδραση. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Το λέω αυτό συχνά στην Ολομέλεια, γιατί όταν έρχομαι στο Κοινοβούλιο, εξακολουθώ ε, να αισθάνομαι μέλο του Κοινοβουλίου. Φυσικά είμαι μέλο τη Επιτροπή τώρα, αλλά νομίζω ότι ήταν καλό σχολείο η μέθοδοι που χρησιμοποίησαμε ε, στο Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό πάντα ζητούσα στην αρχή και έλεγα ότι αφήστε με στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν μεγάλη εμπειρία και δεν θέλω να μετακινηθώ. Αυτό ισχύει για όλη την Επιτροπή. Ο Ζαν Ιούγκερ υποστηρίζει πραγματικά τους στόχους μας και αυτό αναφέρεται και στην επιστολή αποστολής μου. Ήταν πραγματικά γεμάτο το καλάθι. Καταφέραμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα περάσουμε. Γι' αυτό και χαρί σε εσά, γιατί τα 4,5 αυτά χρόνια είσαστε πραγματικά ε, πολύ επικοδομητικοί στη συνεργασία μα. Πάντα είχατε καλέ γραμμέ, πάντα συζητήσαμε τα ζητήματα που μα απασχολούσαν, προετοιμάζαμε του τρομερεί διαλόγου μα και πιστεύω ότι στο ίδιο πνεύμα μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα κάποιο περιθώριο, αλλά ο καιρός ε, τελειώνει. Αύριο συνεχίζουμε με την ε, ισορροπία προσωπικής και εργατικής και επαγγελματικής ζωής. Είναι πολύ τριμερεί διάλογοι που είναι σε εξέλιξη. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν το χρειάζεται να το ακούσετε αυτό, το ξέρετε. Σα ευχαριστώ όμως για την καλή συνεργασία. Καταθέτουμε προτάσεις ε, και αν δεν υπάρχει σωστή αντίδραση, αν δεν υπάρχουν ε, οι σωστές τροπολογίες, δεν θα προχωρήσουμε. Θέλουμε λοιπόν τα καλύτερα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω επίση και τον πρόεδρο τη Επιτροπή, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή συνεργασία. Στο ψητό τώρα. Έγιναν ερώτηση για την ε, πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων. Πώ να αυξήσουμε την απορρόφηση αυτών. Πραγματικά είναι υψηλή η ανεργία των νέων. 6,7% είναι η ανεργία, αλλά πάνω από 14% στους νέου. Έχουμε τρει χώρε με ανεργία των νέων πάνω από 30%. Πολλά λοιπόν απομένουν να γίνουν. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Καταρχάς το πού, πού θα δείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ έχουμε 110 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο που τα κράτη-μέλη που έχουν ποσοστό αναγκών πάνω από το μέσο όρο θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 10% των κονδυλίων ESF για την ανεργία των νέων. Τι κάνουμε για να τα υλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά. Συστάσεις, προτάσεις, κίνητρα. Ομαδοποιούμε τα κράτη-μέλη για να τα αναγκάσουμε να διδαχθούν από τους άλλους. Αυτό πραγματικά που φέρει καρπούς. Και φυσικά αυτό που λέμε είναι ότι θα χρειαστούμε μια ενεργή αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε υπηρεσίες για την αγορά εργασία. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στι συστάσει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι εργαλεία τα οποία χρειάζεστε για να σημειωθεί βελτίωση στο σημαντικό αυτό τομέα. Και να μην ξεχνάμε, γιατί είμαστε και στην Επιτροπή Επασχόληση, ότι χρειαζόμαστε και τι σωστέ μακροοικονομικέ πολιτικέ. Καλό ε, επιχειρηματικό κλίμα για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσει εργασία τελικά οι επιχειρήσει. Ο πυλώνας και πώς ε, μπορούμε να καταστήσουμε το κοινωνικό πύλωνα αρκετά εμφανή στις, ε, στα έγγραφά μας. Έχουμε τις 20 αρχές του πυλώνα. Παρακολουθούμε και με τον πίνακα αποτελεσμάτων το scoreboard αυτό το οποίο έχει ενταχθεί στο εξάμεινο. Έχουμε τις εκθέσεις ανά χώρο και λαμβάνουμε υπόψη τα όσα ε, καταλήγει, στα όσα καταλήγει οι εκθέσεις αναχώρα και καταλήγουμε στα CSR τελικά. Και στην Ευρωζώνη έχουμε πέντε βασικές ε, συστάσεις. Η μία εξ αυτών έχει να κάνει με τις κοινωνικές συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι γίνεται προκειμένου να καταστεί ο πυλώνας αυτός πιο αποτελεσματικό. Αυτό βοηθάει. Και φυσικά την, ε, στην επόμενη φάση και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί φυσικά τα κονδύλια είναι πολύ σημαντικά και υπάρχει στέντρο σύνδεσμο μεταξύ των, του εξαμήνου και των διαφορετικών ταμείων. Αυτό δεν αρέσει στα κρατη Πρέπει να τους το υποδείξουμε με φιλικό τρόπο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι τα πορίσματα στις χώρες μετά από την άσκηση του εξαμήνου με το scoreboard, το κοινωνικό scoreboard κλπ αυτά τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα σχετικά λειτουργικά προγράμματα των ε, ταμείων των κονδυλίων στις συζητήσεις με, την, ε, με τα κρατημέρια. Θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό αυτό σκέλος. Δεν μετρώνουν μόνο τα κοινωνικά ζητήματα και τα δημοσιονομικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και κοιτώντα την ε, δημοσιονομική κατάσταση, την προπολογισμό, όλα τα κρατημέλη είναι κατά το 3%. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι εντελώ διαφορετική προφανώ η εικόνα από τη χρονιά που ξεκίνησε η θητεία μα. καποια κρατημέλη, προφανώ όμω έχουν ακόμα πολλά να κάνουν. Αναλύσαμε τα, τα σχέδια του προπολογισμού, στείλαμε τα σχόλιά μα προ τα κρατημέλη, Συνεχίζεται το εξάμεινο τώρα. Μετά έχουμε τι εκθέσει αναχώρα. χώρα και τέλος τις συστάσεις αναχώρα. Στην παρούσα λοιπόν φάση δεν θα σχολιάσουμε τις μεμονωμένες προτάσεις που έχουν κρατεθεί σε διάφορα κράτη-μέλη. Θέλουμε να κοιτάξουμε το σύνολο της κατάστασης και να κρίνουμε τη σωστή χρονική στιγμή. Για την απασχόληση των νέων δεν μπορούμε να ξεχάσουμε φυσικά ποτέ το σκέλος των προσόντων. Το είπατε πολύ στις παρεμβάσεις σας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι άλλωστε αυτό αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα στους στόχους μας. Ε, η πρόσβαση και στην αγορά αλλά και στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στη διαβίου εκμάθηση και εκπαίδευση. Για την καλύτερη εκτίμηση, αν θέλετε, τη επαγγελματική ε, κατάρτισης και εκπαίδευση να έχουν καλύτερες ευκαιρίες οι νέοι αυτοί και στο πρόγραμμα Erasmus Pro. Έχουν τώρα δυνατότητα ως, ε, όπως και οι πανεπιστημιακοί φοιτητέ να κάνουν ανταλλαγές και να πάνε σε άλλη χώρα. Αυτό θεωρώ ότι δείχνει σεβασμό. Χρειαζόμαστε και πιο πολλούς τέτοιου φοιτητέ. Χρειάζονται να τους σεβόμαστε λοιπόν. Και πιστεύω ότι ήταν αφεντικό το γεγονός ότι όλοι το υποστηρίξαμε. Γιατί τι ανισότητες τώρα. Για το κοινωνικό αυτό scoreboard. Είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσετε για να πείτε στις ε, ε, κυβερνήσεις σας αν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτώντας το S20 και το S18 σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ε, εισοδημάτων ε, σε σχέση με τις πιο πλούσιες χώρες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση σε ό,τι αφορά τις ανισότητες πέρσι. Είμαστε στο 5,2, τώρα είμαστε στο 5,1. Είναι φυσικά ανεπέστατη η αλλαγή. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο προκρίσης. Υπάρχει ακόμα μια διαφορά 0,4%. Είναι πολλό με μεγάλη τη διαφορά. Πρέπει να επιστρέψουμε στα επίπεδα πρώτης κρίσης. Αυτά προφανώ είναι ζητήματα τα οποία συχνά είναι στα χέρια των κρατών μελών. Δεν μπορούμε απλά να νομοθετήσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Τα λαμβάνουμε όμως αυτά υπόψη. Κάνουμε συστάσεις και νομίζω ότι στην παρούσα φάση μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα θέμα αυτό στο οποίο θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Χθε έγινε μια καλή συζήτηση στην Ολομέλεια για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, τι ευκαιρίε για του πολίτε, για του εργαζόμενου. Και νομίζω ότι αν λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζονται για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και την καταπολέμηση των αισθητήτων, Νομίζω ότι με το συνδυασμό αυτών των δύο στόχων βρισκόμαστε σωστό στο δρόμο και αυτό το έθεσε ω ερώτημα και μια πολιτική ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο. Τι κάνουμε τώρα με του ανθρώπου που είναι ηλικιωμένοι. Που δεν έχουν ε, την ε, σωστή εκπαίδευση, τα προσόντα, δεν είχαν ποτέ ε, μια μόνιμη δουλειά. Καταπολεμούμε τον κατακαιρματισμό στα κράτη-μέλη. Η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι οι συστάσεις δεν αποτελούν μόνο ένα κομμάτι χαρτί. Φαίνεται ότι είναι μια σύσταση, ένα πολύ ήπιο εργαλείο, αλλά διαρκώς ζητούμε να μας στέλνουν τα κράτη-μέλη τις στρατηγικές τους, τα σχέδιά τους, τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει μετά από 1,5 χρόνο. Αξιολογούμε λοιπόν τώρα τα έγγραφα που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ε, σχετικές ε, εγγύησεις, την εγγύηση δεξιοτήτων. Άρα εμ, ε, καλούμε τα κράτη-μέλη και παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν πραγματικά κάτι, να αναλάβουν δράση, όχι μόνο να αναφέρουν στοιχεία στο Συμβούλιο και να μένουν στα λόγια. Η εγγύηση για τα παιδιά. Νομίζω ότι η παιδική φτώχεια είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Θα πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Πώς μπορούμε να καταρθίσουμε μια στρατηγική καταπολέμηση του φαινομένου. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική σε βάθος χρόνου. Αλλά φυσικά η φτώχεια των παιδιών σημαίνει ότι υπάρχει φτώχεια στους γονείς. Δεν μπορούμε λοιπόν να εστιαστούμε μόνο στη φτώχεια των παιδιών. Χρειάζεται να παρέχουμε υπηρεσίες στους γονείς, υπηρεσίες που χρειάζονται. Και σε ό,τι αφορά τους γονείς που ε, θέλουν και μπορούν να εργαστούν αλλά δεν έχουν φύλαξη για τα παιδιά τους και γι' αυτό δεν εργάζονται. Όλα αυτά αναφέρονται στις συστάσεις αναχώρα και φυσικά υπάρχουν και τα πρακτικό προγράμματα για ε, την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, διάφορες μελέτε που μας δείχνουν τι μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Έγινε και μια ερώτηση για τη στέγαση. Εδώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι εδώ δεν κάναμε αρκετά πράγματα. Είναι εθνικά, τοπικά, περιφερειακά τα ζητήματα αυτά φυσικά. Κάνουμε συστάσεις, παρατηρήσεις στις ε, συστάσεις αναχώρα σε ό,τι αφορά τις διάφορες φούσκες, τις ε, πολύ υψηλές τιμές, ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. δεν συζητήσαμε παρκώς την άλλη πλευρά του νομίσματος, αυτούς που δεν έχουν στέγαση. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πιο επισταμένως. Δεν είναι προφανώς, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε πλευρά του ευρωπαϊκού επίπεδου τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Η κυρία Αγία έφυγε, δεν χρειάζεται να απαντήσω τι ερωτήσει της φαντάζομαι. Προσπάθησα να επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία, γιατί ξέρω ότι έχετε να ψηφίσετε κιόλα. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε και το μέλλον. Γιατί το μέλλον είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε και ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα. Αλλάζουν οι αγορές εργασίας, οι δεξιότητες που αυτή τη στιγμή χρειάζονται στην αγορά εργασίας, αλλάζουν και αυτές. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτό προβλέπει άλλωστε και ατζέντα και το πανόραμα για τις επαγγελματικέ δεξιότητες και τα σχέδια που συνενώνουν και συγχωνεύουν, αν θέλετε, και τομείς, αλλά και πανεπιστήμια, εργοδότες, εργαζόμενους, συνδικαλιστές, για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες. Ποιες είναι οι ανάγκες που θεωρούμε ότι υπάρχουν και που θα καθοδηγήσουν την ε, με την ε, εκ νέου εκπαίδευση ατόμων. Θα πρέπει να γνωρίσουμε επίση τι δεξιότητε οι οποίε αποκτώνται στα πλαίσια τη ανεπίσημη ε, εκπαίδευση και κατάρτιση και αυτό είναι στόχο τη ατζέντα και σε αυτό πραγματικά καταβαλούν προσπάθειε και τα κράτη-μέλη. Ε, ακούσαμε και κάποια στοιχεία για την φορολογική πολιτική. Φυσικά. Υπάρχει ε, η κοινωνική νομοθεσία, το κοινωνικό ταμείο, η συνεργασία στα πλαίσια του εξαμήνου. Αυτό ισχύει και σε άλλες πολιτικές. Όταν δεν υπάρχει δική φορολόγηση, πώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη, πώς μπορούμε... Αν δεν σεβόμαστε του κανόνε ανταγωνισμού, πώς μπορούμε να πούμε ότι ζούμε σε ένα δίκαιο κόσμο, αν δεν ε, υπάρχει κάποια αντίδραση όταν υπάρχει ε, διακριτική μεταχείριση σε κάποια κρατημέλη ορισμένων επιχειρήσεων ει βάρο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποτελούν αδικίες. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε στην Επιτροπή μας και η Επιτροπή Φεστάγκεν που αναφέρατε και από πλευρά του Επιτρόπου Μοσκόπηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Το CCTV, το ψηφιακό φόρο είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα. Τα αναφέρω ενδεκτικά. Στην πτυχή του φίλου. Πάντα ζητώ. Να αναφέρετε το θέμα αυτό όπου μπορείτε. Το διαπιστώνουμε ξανά και ξανά στον τομέα της ε, απασχόλησης. Αυξήθηκε κάπως το ποσοστό απασχολησιμότητας και απασχόληση των γυναικών, αλλά υπάρχει ακόμα χάσμα. νου είσαστε εισηγητής, ε, εισηγήτρια για την Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και είσαστε υπεύθυνοι για την έκθεση για την ισορροπία επαγγελματική και προσωπικής ζωής. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν δίκαιη κατανομή των ε, καθηκόντων μεταξύ γυναικών και ανδρών και στα πλαίσια της οικογένειας και στα πλαίσια της εργασίας και θεωρώ ότι αυτή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική προσωπική ζωή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τα μακροοικονομικά στοιχεία. Το χρειαζόμαστε το στοιχείο αυτό και τι περιφέρειε. Δύσκολο και αυτό. Ζω σε ένα κράτο μέλο με υποσπονδιακό χαρακτήρα. Έχουμε μόνο τρει περιφέρειε και ήδη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με τι τρει αυτέ περιφέρειε. Γιατί υπάρχουν διαφορέ, υπάρχουν διαφορετικέ ε, προτιμήσει αυτό δεν αρέσει συχνά στον κόσμο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε κάθε περίπτωση θα έχουμε συνομιλία με όλες τις περιφέρειες στα πλαίσια του εξαμήνου. Έχουμε 230, αν δεν κάνω λάθος, περιφέρειες στην Ευρώπη. Πώς θα τις προλάβουμε όλες. Όταν όμως κάνουμε τις εκθέσεις αναχώρα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό το γεγονό. Μπορούμε να μιλάμε για τα ποσοστά ανεργία για ένα κράτο μέλο, αλλά αυτό ενδεχομένω να διαφέρει τόσο δραματικά από το βορρά στο νότο, χρειάζονται τα στοιχεία αυτά. Χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και αυτό δεν είναι πάντα σαφές σε όλες τις εκθέσεις, γιατί είναι ουσιαστικά αδύνατον να ολοκληρωθεί στην περίπτωση αυτή η άσκηση. Το έχω όμως υπόψη μου. Το χάσμα και το κενό, οι διαφορές που υπάρχουν στις, ε, στους μισθούς για τους κοινωνικούς εταίρους, για τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι φατικό το ότι το ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι στην παρούσα φάση. Αυτό. Και το συζητιέται το θέμα αυτό και μεταξύ των κρατών μελών. Και βλέπουμε ότι αυτό καθίσταται όλο και πιο σημαντικό. Μακροπρόθεσμη ενεργεία και το... Εδώ θα κλείσω. Η μακροπρόθεσμη ενεργεία σε βάθος χρόνου τέτοια μειώνεται. Αυτό είναι καλή είδηση από 4% 3,4% φέτος. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά ακόμα πολλά έχουν να γίνουν. Γιατί υπάρχουν κρατημέλη που είναι στο 1,9% και άλλα κρατημέλη είναι στο 17% σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη ενεργεία. Μεγάλες διαφορές λοιπόν. Αυτά, Πρόεδρε, γιατί πρέπει να φύγετε κιόλα. Ναι, πρέπει. Πρέπει, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, σας ζητώ μόνο να με βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε και εμείς εσάς για να ολοκληρώσουμε τα θέματα που έχουμε, να τα φέρουμε σε αίσιο πέρας. Αλλά να μην ε, προσπαθήσουμε να έχουμε το καλύτερο και τελικά δεν έχουμε τίποτα. Ξέρουμε, πώς το λέμε, το, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού, κάπως έτσι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να μην ε, επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή λύση χωρίς συμβιβασμούς, γιατί στο τέλος θα μείνουμε με αδία Να ολοκληρωθούν τριμερείς διάλογοι, υπάρχουν μερικοί ακόμα και χρόνο έχουμε μόνο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου περίπου, δηλαδή. Δεν τελειώνει ο χρόνος μας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και πάλι και τα ανταποδίδω. Με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα μαζί σας και θα συνεχίσουμε και το 19. Καλές γιορτές σε όλους. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τέισεν. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Αλλά έχουμε πάρει τροφή για σκέψη για τα Χριστούγεννα. όλοι. Έχουμε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Α, μάλλον κάτι φανταστικό που μπορούμε να ζούμε ως εμπειρία. Γύρισε ο κύριος Χέντελ. Του δίνω το λόγο για να μας πει μερικά λόγια, παρακαλώ. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι ξαναγύρισα Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ειλικρινά, όλους εσάς που μου στέλνετε τους χαιρετισμού κατά τη μακρά διάρκεια της ασθένειάς μου. 12 εγχειρήσει έκανα, αλλά ήξερα πάντα ότι ήθελα να επιστρέψω εδώ, να είμαι στο πλευρό της Μαριάν Τάισεν και της Μαρίτα Ουλφσκοκ για να ολοκληρώσω εδώ το έργο που είχα να κάνω στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Πολλοί από σας μου έστελαν χαιρετισμού, ευχέ, κάρτε. Ε, ήσασταν στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά. Ήταν δύσκολο το διάστημα αυτό. Αλλά νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο για να επιστρέψω θα χρειαστεί κάποιο καιρό για να ξαναβρω τη φυσική μου κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μπορώ να είμαι εδώ για να αγωνιστούμε το τελευταίο διάστημα μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πρόεδρος. Πραγματικά ζούμε μια φανταστική εποχή που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ θαυμαστά πράγματα και στην πολιτική και στην οικονομία αλλά και στην υγεία. Ε, έχω μια ε, κόρη που είναι ογκολόγος και μου είπε ότι σήμερα όλα είναι δυνατά, σχεδόν τα πάντα. Δεν μας εκπλήσει τόσο πολύ, αλλά νιώσατε τη ζεστασιά των συναδέλφων. Την ευχαρίστα, την Επίτροπο νομίζω ναι. Ε, και τώρα ε, έχετε το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα το επαναλάβω, θα πέρασουμε στο τελευταίο θέμα ε, στην ημέρη σε διάταξη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Οικονομικό Συντονισμό και θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάρκιν που μάλλον κάποια στιγμή θα έρθει να μας παρουσιάσει το θέμα της το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής για την ετήσια ανάπτυξη το 2019. Έχετε το λόγο κυρία Χάρκη. Έχουμε μείνει λίγοι ελεκλεκτοί και θα σας ακούσουμε προσεκτικά. Για σύντομη παρουσίαση γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Χάντλ, καλώς ήρθατε. Χάντλ, καλώς ήρθατε και πάλι. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη συζήτηση το έχουμε ήδη κάνει σήμερα το πρωί. Πριν πω λοιπόν, έχω αντί να μπω σε λεπτομέρειε για τα θέματα αυτά, πολύ σύντομα θα σα δώσω μερικά σημαντικά σημεία που τα αφορούν. Ξεκινώ λέγοντα ότι όλη η εικόνα μου φαίνεται θετική. Ε, οι κύριες τιμές, ε, οι κύριοι δείκτες φαίνεται να πηγαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο κάποια στοιχεία βλέπουμε, εάν κοιτάξουμε πιο λεπτομερώς, ότι παρουσιάζουν και κενά. Και εδώ στην έκθεσή μου, που είναι αναγκαστικά πολύ σύντομη και ελπίζω να υπάρξουν πρωτοβουλίες, ε, μετροπολογίες οι οποίες θα τη συμπληρώσουν και θα τη βελτιώσουν. Ε, κάποια λοιπόν από τα σημεία που εγώ ε, τονίζω είναι ο κίνδυνος της φτώχειας. Αυτό που συζητήσαμε και σήμερα το πώς μπορεί το εξάμεινο να αξιοποιηθεί για την εξέβρεση λύσεων και είπε και η συνάδελφος Ρομπέρο νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να προσπαθήσουμε να ε, τιμωρούμε τα κράτη-μέλη, αλλά να τα ενθαρρύνουμε ώστε η καταπολέμηση της φτώχειας να, είναι, να γίνει πραγματική προτεραιότητα για αυτά. Μας είπε η Επιτροπή 1 και 5 όταν μιλούμε για κοινωνική και οικονομική πολιτική. Εγώ νομίζω πρέπει να φτάσουμε στο 2 και 5. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέους τρόπους και ρύθμιση των, ε, των νέων μορφών εργασίας ε, και εξασφάλισης πρόσβασης χωρίς να επεκταθώ σε αυτά, θα σταματήσω σε αυτό, ε, σε αυτό το σημείο για να πάω στο, σε εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο, που είναι το εισόδημα των οικοκυριών. Αυτό παρουσιάζει πολύ πιο βραδία από το ΑΕΠ ανάπτυξη και ενώ ξέρουμε ότι είναι τελείως άνηση η κατανομή των εισοδημάτων χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χειρότερη. Έχουμε ένα μεγάλο χάσμα λοιπόν το οποίο συνεχίζεται έστω πιο αργά από τις άλλες χώρες αλλά δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε να συνεχίσει να αυξάνεται και είναι από τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε και η στέγη αναφέρθηκε τεράστια κρίση σε πολλέ χώρες και στη δική μου πρέπει να βρούμε λύσεις για το πώ θα μπορεί κανεί να πληρώνει ένα κατάλληλο ε, και να έχει και πρόσβαση σε μια κατάλληλη στέγη. Το ότι δεν υπάρχει κοινωνική στέγη. Βέβαια, η Επίτροπο μα είπε: Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ. Αλλά από την άλλη, μιλούμε εδώ για κοινωνικέ επενδύσει. Γιατί να μην προσπαθήσουμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο από κοινού, δημοκρατική αλλαγή, συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, στέγη που να μπορεί να αντέξει το βαλάντιο του μέσου πολίτη και έχουμε πρόβλημα ε, όχι απλώς λόγω του χάσματος στον πλούτο ή των ανισοτήτων στον πλούτο, αλλά και των ανισοτήτων και των ελλείψεων σε επενδύσεις. Αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Οι μακροπρόθεσμα άνεργοι επίσης χρειάζονται πολύ πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα με βάση τα όσα μας προσφέρει σαν δυνατότητα και το Ταμείο για την των Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης, αλλά και την εμπειρία που έχουμε συλλέψει μέχρι στιγμής. και πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βρουν ε, κάποιες λύσεις. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ε, ανεργία των νέων 10% που τα συστήσαμε και με την Επίτροπο νωρίτερα. Καλό είναι αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο, δεν φτάνει. Επίσης, άτομα με αναπηρία υποστήριξη μικρομεσαίων, ε, φτώχεια των παιδιών, έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, πολλά είπα ήδη, πολλά άλλα θα μπορούσα να πω, αλλά θα σταματήσω περιμένοντας τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Η Σκιώδης παρακαλώ. Κυρία Κοζλόφσκα. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. που είστε εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ κύριε Χέντελ μαζί μας. Ε, εξαιρετικό το ότι σας βλέπω πάλι κοντά μας. Για την έκθεση ευχαριστώ και συγχαίρω την κυρία Χάρκιν. για την κοινωνική ευαισθησία που δείχνει, για την ισότιμη ε, με κατανομή των ε, εισοδημάτων ε, και του πλούτου. Θα ήθελα κάποιες μικρές τροπολογίες να προσθέσω, οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με τη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά της εργασίας, θα έχουν κάπως περιορισμένο δηλαδή πεδίο και την επιδίωξη μιας δικαιοσύνης κοινωνικής μέσω της συμμετοχής της γυναίκας στο εργασιακό γίγνεσθε. Πολλές άλλωστε είναι οι γυναίκες ε, που εργάζονται χωρίς κοινωνική ασφάλιση και αυτό αφορά περισσότερο το τομέα της μέρημνας ε, για το με ανάγκες ε, της πρόνοιας δηλαδή της κοινωνικής, πράγμα το οποίο βεβαίως επηρεάζει γενικά τα, το, την κοινωνική τους προστασία και πάνω απ' όλα τα εξωτικά τους δικαιώματα. Σε αυτό θα αναφερθούν οι προστορέ μου τροπολογίες. Θα μιλήσω επίσης για τομεί το, ε, ελληματικούς ως προς ε, καταρτισμένο προσωπικό, ε, ενίσχυση της επαγγελματική και πρακτικής κατάρτισης, ε, κινητικότητα, βασικές δεξιότητες, που είναι πολύ σημαντικό, το αναφέρετε και εσείς με το 20% της του λειτουργικού αναλφαβητισμού ε, ή παράγωγου αναλφαβητισμού όπως λέμε στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί δηλαδή εκτός από τα basic skills ή μάλλον στα basic skills πρέπει να περιλάβουμε και τις ψηφιακές δεξιότητες γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε σε μια πραγματικά καινοτόμο ε, οικονομία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Γανά έχει φύγει. Κυρία Τρεμπέσιος, επίσης, Γκουέντζιέλ Κάνες η κυρία Λάμπερτ. Είναι εξαιρετική, εξαιρετικά καλή βάση έκθεση της ε, συναδελφού ε, Χάρκιν η έκθεση αυτή. Τα είπα τα βασικά σχόλια στη συνομιλία με την Επίτροπο. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ορισμένα ζητήματα, το ζήτημα της στέγης, το τονίζω περισσότερο, ε, κάποια από τα σημεία του αρχικού κειμένου της Επιτροπής που έχουν να κάνουν με τη χρηστή διακυβέρνηση, ε, την επικοινωνία με τον πολίτη ουσιαστικά γιατί πολλές φορές ο δεν γνωρίζει τι δικαιώματα έχει για να τα διεκδικήσει περιβαλλοντική πτυχή βεβαίω που θέλουμε επίση να αναδειχθεί περισσότερο. Αλλά πάντω είναι καλή βάση, πολύ καλή βάση για... και θα δουλέψουμε πάνω Αλλά μετά τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Έχω ξεχάσει κανέναν. Να. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κυρία Χάρκιν. Όχι, ευχαριστώ του συναδέλφου μόνο. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Προθεσμία για τροπολογίες μόνο στα αγγλικά 9 Ιανουαρίου το μεσημέρι στις 12. 26 με 27 η συνεδρία στην οποία θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και μετά ολομέλεια το Μάρτιο. Αυτά ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε όλο να σας ε, πιέζω και ορισμένοι τόσο πολύ απογοητεύτηκαν που έφυγαν εν τέλει, αλλά τα καταφέραμε, τελειώσαμε και έχουμε και ένα περιθώριο 5 λεπτών μέχρι να πάμε στην Ολομέλεια για τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά.